διαδικαστικής παρέμβασης του κύριου Κόρβετ. Κύριε Κόρβετ, έχετε το λόγο. Δεν μας είπατε τίποτα για αποχώρηση βουλευτή, ο οποίος αποχωρεί από κάποια βουλευτική ομάδα. Σας το λέω αυτό γιατί το UKIP δημιούργησε ολόκληρο επεισόδιο σχέση με κύριε Άνιστον η οποία ε, απευλήθη του κόμματος αυτού. Όμως εδώ παραμένει μέλος της ε, πολιτικής ομάδας εγκρυπτό και απαραβίστο έχει παραμείνει εδώ και αυτό το κάνουν τόσο ώστε μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα τα οικονομικά τα οποία προβλέπεται να χορηγούνται προς την πολιτική ομάδα. Αυτό δεν είναι ευχαριστασμός και υποκρισία ή, απλώ απλώς δεν τα είπαν σωστά. Κύριε Κόρμπετ, μια στιγμή. Μια στιγμή λέει ο πρόεδρος. Καθίστε, θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Κόρμπετ. Είστε ένας πεπειραμένος συνάδελφος. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το άρθρο της ημερής του κανονισμού μας επί του οποίου εδράζεται η διαδικαστική σας παρέμβαση. Αν μου λέγατε ποιο άρθρο θα ήταν αυτό, θα μπορούσα να αναφερθώ για το θέμα αυτό. Δεν είπατε τίποτα όμως για το άρθρο του κανονισμού. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο σε αυτά που λέτε. Δύο πράγματα θέλω να επισημάνω. Εσείς ξέρετε ότι οι αποφάσεις για την παρουσία βουλευτών σε μια κοινοβουλευτική ομάδα δεν παίρνονται από τα πολιτικά κόμματα τα ηχεία στις χώρες μέλη, αλλά από τις ίδιες πολιτικές ομάδες εδώ. Επομένως αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί σε συζήτηση ή σε πληροφόρηση τη ολομέλεια. Δεύτερον, υπάρχει μια παραβίαση κανόνων από τη δική σα πλευρά που δεν, είναι αποδεκτή. Κύριε Ντάρτμου, θα έχετε το λόγο. Just simply Απλώς σας αναφέρω το εξής. Είναι θέμα νομικό και διαδικαστικό. Αλλά είναι και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τόσο σας ενδιαφέρουν. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται και ο κύριος Κόρμπετ ε, για αυτά βέβαια. Γιατί η συνάδελφος ενεργεί μέσω αντικλείδου της δικηγόρου. Και παραμείνει στο κόμμα δυνάμει του κανονισμού του Κοινοβουλίου και του ιστορικού μας κανονισμού και θα συνεχίσει. Δεν ξέρω ε, μήπως έτσι σας καθησύγασε κύριε Κόρμπετ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, αλλά και η δική σας παρέμβαση δεν έχει καμία σχέση με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου και δεν είναι διαδικαστική παρέμβαση. Κύριε Μπορέλη. Για την ευθυντή θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Τελείσε αναστολή η συνάδελφος αυτή. Μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι αστυνομικές έρευνες και να ληφθεί η οριστική απόφαση της πολιτικής ομάδας. Αυτό ήταν μια απάντηση που συνάδει με τον κανονισμό στην ερώτηση του κυρίου Κόρμπετ, κύριε Μπορέλη. Ευχαριστώ. Βάσει του άρθρου 149 ε, η επίσημη, το επίσημο σχέδιο της ε, ημερήσιας διάταξης έχει διανεμηθεί. Προτείνω μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη την ε, δήλωση της Κομισιόν για την πυρκαγιά στο, στο εργοστάσιο του Μπαρκαντές και το σύμφωνο βιωσιμότητας με τον Μπακλαντές να εξεταστεί σε μια μεταγενέστερη συνεδρίαση. Υπάρχουν αντίρρηση σχετικά ούτως απεφασίστη. Κύριε Γκόλης, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Διότι είδαμε τις καταστροφές της παγκοσμιοποίησης του διεθνούς καπιταλισμού του κοινικότερου είδους που επωφελείται από τους χαμηλούς μισθούς εκείνων που εργάζονται σε απαράδεκτες συνθήκες δουλείας σχεδόν. Τα προϊόντα τους έρχονται χωρίς δασμούς να καταστρέψουν τις δικές μας επιχειρήσεις και βιομηχανίες και εκτός αυτού θεωρώ ότι η πολιτική αυτή ευθύνεται για εκατοντάδες θανάτους και εμείς οι Ευρωπαίοι και οι Δυτικοί είμαστε συλλογικά αν και έμεσα συνυπεύθυνοι και γι' αυτό νομίζω ότι το σχέδιο αυτό δεν πρέπει να πρέπει να αφαιρεθεί από την κοινωνική διάταξη αμέσως. Ευχαριστούμε κύριε Γκόλνης. Είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες ζήτησαν την ε, αναβολή αυτού του σημείου. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν ποιοι υποστηρίζουν την ε, αναβολή της συζήτησης για το θέμα του Μπαγκλαντές. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια πλειοψηφία για την αναβολή. Κύριε Γκόλης, έχετε και πάλι Η ομάδα σας ζήτησε η ομάδα του ΕΡΚ ζήτησε να προσθεθεί μια συζήτηση για την ε, αντίλωση Κομισιόν σε σχέση με τη συμφωνία PNR με το Μεξικό να προσθεθεί ως δεύτερο σημείο μετά από τις ε, ε ψηφοφορίες. Επομένως η συνεδρία μας θα συνεχιστεί μέχρι τις 10 η ώρα. Η κυρία Χόλμαϊερ θέλει να κάνει μια παρέμβαση σε σχέση με το θέμα αυτό. Παρακαλώ κυρία Χολμάιερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αίτησή μας είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι το Μεξικό έχει θέσει μια προθεσμία καταληκτική σε σχέση με, τις, ε, με τα πρόστιμα τα οποία θα τεθούν εάν δεν δίδουν αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση ώστε να μην εφαρμοστούν όλα αυτά τα πρόστιμα, να υπάρξει μια συμφωνία μέχρι τις 30 Ιουλίου. Θα ήθελα να ξέρω από την Κομισιόν τι θα γίνει μέχρι την ημερομηνία αυτή. Η κυρία Ινφέλτ θέλει να λάβει το λόγο σχετικά. Χωρίς μικρόφωνο. Έχω υποβάλει έτοιμα επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια από το αυτό να μπει στη μέσα σε διάταξη. Οπότε βεβαίω και είμαστε υπέρ του αιτήματο πάντω. Α αλλάξει ελαφρώ ο τίτλο. Γιατί είναι ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σύναψη τη συμφωνία. Πρόκειται για σχέδιο συμφωνία. Οπότε είμαστε υπέρ της ε, αναβολής και θέλουμε να υπάρξει τροποποίηση του τίτλου. Κάποιος θέλει να αναφερθεί κατά της ε, αίτησης αυτής. Όχι. Προτείνω στην κυρία Χολμάιερ και την κυρία Ινφέλτ να, να πούμε ε, ότι είναι μια συζήτηση για την προτινόμενη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μεξικό για το PNR. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης κυρίας Χόλμαιερ θα σηκώσει το χέρι του παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Η αίτηση αυτή γίνεται δεκτή λοιπόν. υπάρχει μια αίτηση των πρασίνων να γίνει μια συζήτηση σε σχέση με τη δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν σε σχέση με την Ελλάδα να εγγραφεί στην δημόσια ε, διάταξη με τίτλο ε, «Εργασίες της Ευρωομάδος και συνέχιση του προγράμματος χωρίς ψήφισμα». Η κυρία Χάρμς έχει το λόγο για να αιτιολογήσει αυτή την αίτηση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουμε αυτές τις λεγόμενες μικροσυνόδους που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επίκαιρα θέματα και εξελίξεις. Όπως βλέπω, τα μέσα ενημέρωσης και τον τύπο στην Ευρώπη είναι σαφές ότι η λέξη Brexit βρίσκεται στα χείλη όλων. Αυτό αναφέρεται και από ανώνυμες πηγές από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή της ευρωπαϊκής κυβέρνησης που δίνουν την εντύπωση ότι το καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το καλύτερο για την Ελλάδα θα ήταν το λεγόμενο Brexit. Αυτό νομίζω ότι αυτό είναι μια πράξη αδράνειας και αμέλειας έναντι των πολιτών μας, έναντι της Ελλάδος. Γιατί αυτό το Brexit θα οδηγήσει σε μια ακόμα πιο σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση για τους πολίτες της, Ευρώπη, της Ελλάδος οι οποίοι έχουν πληγεί από έτη οικονομικής κρίσης. Πιστεύω ότι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο η Ευρωζώνη σε οικονομικό επίπεδο, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να εκτεθεί σε ένα τεράστιο κίνδυνο αν επιτρέψει να συνεχιστεί αυτή η σπερμολογία σε σχέση με το Brexit. Πιστεύω λοιπόν ότι το κοινοβούλιο μας, το οποίο είναι ο χώρος συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει ακριβώς σε αυτή τη χρονική στιγμή να συζητήσει για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Έχετε την προσοχή μου, αλλά ίσως δεν έχετε την προσοχή άλλων συναδέλφων. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης, κύριε Χάμς. Μάλλον, αν θέλει κάποιος να λάβει το λόγο υπέρ αυτής της πρότασης. <clears throat> Θέλετε να μιλήσετε, κύριε Λούκε. Αυτό με εκπλήσει κύριε Λούκε που θα υποστηρίξετε την πρόταση της κυρίας Χάμς. <coughs> Σας ευχαριστώ που μπορώ εγώ από μόνος μου να αποφασίσω τι θα πω και τι δεν θα πω. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η πρόταση της κυρίας Χάμ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιληφθεί κατεπηγόντως για το θέμα αυτό, γιατί η επίσημη θέση <coughs> της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει αναφερθεί από τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης, μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ε, κανένα Brexit. Είναι αδιανόητο μια χώρα να βγει από την Ευρωζώνη. Το έχει πει, το έχει γράψει η Κομισιόν, αυτή είναι η επίσημη θέση, αλλά αυτή τη στιγμή <clears throat> υπάρχουν πολλοί ε, αναλυτές, μελετητές και μέλη κυβερνήσεων ακόμα που έχουν αναφερθεί στο θέμα του Brexit. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Κομισιόν. Θα υποστηρίξει κάποιο Brexit. Υπάρχουν προετοιμασίες για κάτι τέτοιο ή είναι άποψη Κομισιόν το Brexit είναι απόλυτα αδύνατο και θα αν τα πράγματα προχωρήσουν έτσι, ίσως κάποια μέρα θα πρέπει η Ελλάδα να φύγει με απόλυτα ε, ανεξέλεγκτο τρόπο από την Ευρωζώνη. Κύριε Λούκε, ήταν κάπως παράξενη αυτή η σύνδεση που κάνετε κύριε Λούκε. Εγώ δεν ήθελα να πω αυτά τα οποία θα λέγατε εσείς. Έχετε κάθε δικαίωμα να πείτε αυτά τα οποία θέλετε. Αντίθετα, εναντίον αυτή τη αίτηση θέλει να λάβει το λόγο η κυρία Τσίμα. Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μου είναι εναντίον αυτή τη αίτηση να γίνει σήμερα μια συζήτηση για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωζώνης και της Ελλάδος γιατί πρώτα απ' όλα πιστεύουμε ότι στις 20 Φεβρουαρίου έχει τεθεί μια βάση για τις διαπραγματεύσεις εργασίας μεταξύ της Ευρωζώνης και της Ευρώπης, εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα αυτή η βάση. Όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν είναι ειδήσει από εφημερίδες, είναι φήμες, έχουμε όμως και πηγές καλά πληροφορημένες όπως είναι η Κομισιόν που συνέχεια διαψεύδονται. Εγώ δεν ξέρω με ποια βάση μπορούμε τώρα να συζητήσουμε. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η φήμη. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για την Ελλάδα, αλλά αυτή πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη. Θα ήθελα να γίνει στην επόμενη μας συνεδρίαση ολομέλες, αλλά κυρίως να αποφύγουμε να γίνουμε κι εμείς υποχείρια φημών που μπορούν να οξύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει σε αυτήν την τωρινή στιγμή και πιστεύω απόλυτα όπως και η κυρία Χάμς, ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι έσχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όνειδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση της κυρίας Χάμς τίθεται σε ψηφοφορία. Ποιος υποστηρίζει την πρόταση της κυρίας Χάμς. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απολύπτεται η έτσι της κυρίας Χάμς. Έχουμε λοιπόν οριστικοποιήσει το σχέδιο εργασιών για σήμερα.